Κυρίε και κύριοι, σα ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σα εδώ. Καθίστε για να μην καθυστερούμε πολύ, γιατί μα πιέζει πάρα πολύ ο χρόνο. Ε, θα ακούσουμε τι ανακοινώσει τη Προεδρία και επειδή έχει πολύ καιρό που δεν ακούσατε τη φωνή του επικεφαλή της γραμματέας, του κ. Λαμπρέ, θα σα πω ότι θα σα κάνει αυτό τι ανακοινώσει. Έχθε στη συνεδρίαση των συντονιστών ελήφθησαν εξή αποφάσεις ε, προ ενημέρωσή σα. Ο κύριο Βόμποντα, ω πρόεδρο, ε, θα συντάξει δύο εκθέσει ε, για την κύρωση και την προσχώρηση των κρατών μελών στη Διεθνή Σύμβαση για την απόδοση ευθύνη και την αποζημίωση για ζημίες για τις ζημιογόνες ουσίε και ρηπογόνε ουσίε από θάλασσα. Η ετήσια έκθεση για το 2014 για την επικουρικότητα και την αναλογικότητα ανατώθηκε. Ο κύριος Τζαμπάνκι θα εκπονήσει έκθεση για την ενιαία μορφή των θεωρήσεων διαβατηρίων και επιπλέον θα υπάρξει ένα ε, εργαστήριο με τη συμμετοχή της Επιτροπής Αναφορών τον Οκτώβριο για τις ε, διεθνείς ε, μειώσεις και θα υπάρξει και ε, προφορική ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο. Θα χρειαστούμε και έναν ακόμα για την αποστολή στην Ουκρανία που θα γίνει στις 24 και 25 Σεπτεμβρίου. Οι συνεδριάση του 2016 θα σας διανεμηθούν ε, σύντομα και τέλος ε, θα ζητήσουμε έγκριση για να εφαρμοστεί το άρθρο 54 για την έκθεση για την εκπροσώπηση των εργαζομένων σε επίπεδο Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Απασχόλησης. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε διότι ε, προσθέσατε λίγη ποικιλία στην ε, μονοτονία των αποφάσεων. Τώρα να δώσουμε το λόγο στην κυρία Λίδια Γκέργεν Δεότεμπερ για την έκθεσή της. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσω πολωνικά από εδώ και πέρα. Χαίρομαι που μπορούμε επιτέλους να ολοκληρώσουμε με την υπόθεση αυτή σήμερα για την, ε, ε, επίλυση των μικροδιαφορών. Πρόκειται για διασυνοριακές ε, μικροδιαφορές την τελευταία φορά σας έδωσα κάποιες πληροφορίες για τον ε, τριμερή διάλογο, ο οποίος ήταν ιδιαίτερα επιτυχής και σήμερα θα ψηφίσουμε. Αμέσως μετά τη συνεδρίασή μας ε, ε, στον τριμερή διάλογο η Προεδρία ακολούθησε τη διαδικασία, υπήρξε και ομόφωνη απόφαση στο Συμβούλιο, χαίρομαι ιδιαίτερα γι' αυτό και νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι με την έκθεση αυτή καταφέραμε να έχουμε κάποιους εξαιρετικούς συμβιβασμούς και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον κύριο Μπούντα ιδίω για την εξαιρετική του συνεργασία, πολύ δημιουργική μάλιστα συνεργασία και θα ήθελα να ευχαριστήσω και όλους τους βοηθούς και τους συμβούλους μας ε, οι οποίοι συμμετέσχουν ενεργά στην ε, εκπόνηση της έκθεσης και θα ήθελα να ευχαριστήσω και εσάς για την αποτελεσματική σας ε, συνεργασία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τη γραμματεία. Ο Άλεξ ε, ήταν παρόν και θα ήθελα να ευχαριστήσω και αυτόν ε, για την εξαιρετική συνεργασία. Και τώρα θα ήθελα να ρωτήσω το εξή. Θα ήθελα να ψηφίσουμε και να υποστηρίξουμε αυτή την πρωτοβουλία, η οποία θεωρείται και από πλευρά μα αλλά και από πλευρά Συμβουλίου μια ιδιαίτερα επιτυχής συμβαστική πρόταση. Ευχαριστώ. C'est d'une rapidité euh, formidable. Ταχύτατα. Αγαπητοί συνάδελφοι, ας ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, έκθεση Γκέριγκερ de Edinburgh. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Εψήφισαν όλοι πέρα στις ψηφοφορίες. Βλέπετε την αποδοχή δημοσκοπικά, έστω και σε δημοκρατίες. Κάνει καλό αυτή η επικρότηση. Λοιπόν, τώρα έχουμε την έκθεση Ντελβουά, δίνω το λόγο στην συνάδελφο αμέσω. Εφόσον βεβαίως σταματήσουν τα σούσουρα και οι ψήφοι στο πίσω τη αίθουσα. Κυρίες μου, παρακαλώ. Ωραίες οι φωνούλες σας, αλλά σα ακούμε μέχρι εδώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Εδώ έχουμε να κάνουμε τον κανονισμό τον σχετικό με τη διευκόλυνση ελεύθερης κυκλοφορίας σε σχέση με την αποδοχή ορισμένων δημοσίων εγγράφων. Θα γνωρίζετε ότι πρόκειται για μια πρόταση της, Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το 2013. Καταργείται η σφραγίδα της Χάγης και η υποχρέωση για την επικύρωση ορισμένων εγγράφων για υποθέσεις πολιτικών για φυσικά πρόσωπα δηλαδή, αλλά και για το καθεστώς και την ε, εκπροσώπηση νομικού προσώπου. Ε, διευκολύνεται η μετάφραση όταν παρουσιάζεται και το πρωτότυπο δεν χρειάζεται επιστοποιημένη μετάφραση. Τρίτον, διευκολύνεται η εισαγωγή, μάλλον εισάγονται πολύγλωσσα έντυπα που αντικαθιστούν τα εθνικά αντίστοιχα και τέταρτον ενισχύεται η συνεργασία μεταξύ κρατών μελών στο σύστημα ημίν που είναι το Internal Market Information System, ε, σύστημα πληροφοριών εσωτερικής αγοράς. Εδώ λοιπόν είχαμε μία πρόταση που υιοθετήθηκε το 2014 με την έκθεση RAPCAI, που είχε επεξεργαστεί την έκθεση αλλά τώρα δεν, έχει, δεν είναι πλέον μελών του Κοινοβουλίου. Γνωμοδότηση με την οποία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε διευρύνει το πεδίο εφαρμογής εισάγοντας και άλλα έντυπα στην, στα όσα έχει αρχικά προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ιδιαίτερα σε θέματα πνευματικής ε, ιδιοκτησίας, σε θέματα ακινήτων, φορολογία, δίπλωματα, ε, πτυχία και ενδεικτικά, σχολικά διευκολύνεται ακόμη περισσότερο η μετάφραση, δεν χρειάζεται πιστοποιημένο αντίγραφο και εφόσον το κράτος το οποίο λαμβάνει ένα έγγραφο είχε αμφιβολίες θα όφιλε εκείνο να ζητήσει τη μετάφραση από το κράτος προελεύσεως του εγγράφου και θα έπρεπε η αρχή που ζητεί τη μετάφραση να καταβάλει και τη σχετική δαπάνη ε, και εισάγονταν πολλά πολύγλωσσα έντυπα. Το Συμβούλιο επί έτη δύο συζήτησε τον κανονισμό αυτών, περιορισμένης εμβέλειας ε, που όμως θα μπορούσε να αλλάξει σοβαρά τη ζωή των πολιτών που ε, μεταβάλλουν την κατοικία τους, μεταφέρουν την κατοικία τους και τώρα έχουμε τις τελικές προτάσεις του Συμβουλίου που συμφωνεί με την κατάρριξη της φραγίδας της Χάγης στο ιστορικό της Ένωσης, αλλά τη διατηρεί στη σχέση με τρίτα κράτη. Λογικό μου φαίνεται. Πολίτης ο οποίος ήδη διαθέτει τη φραγίδα της Χάγης μπορεί να τη χρησιμοποιήσει, άρα μπορεί να υπάρξει μια συνύπαρξη του νέου συστήματος με την σφραγίδα της Χάγης, αλλά θα πρέπει να ενημερώνεται ο πολίτης ότι δεν ε, υποχρεούται πλέον να χρησιμοποιεί τη σφραγίδα της Χάγης. Επίσης περιορίζει το πεδίο εφαρμογής για άλλη μια φορά το Συμβούλιο, δηλαδή αφορά μόνο ζητήματα του αστικού δικαίου και συγκεκριμένα της οικογενειακής κατάστασης, άρα αφορά μόνο τους πολίτες και όχι τις, ε, τα νομικά πρόσωπα, η αλλαγή αυτή, ορισμένα μόνο έγγραφα δηλαδή υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής, άρα πρόκειται για γέννηση, θάνατο, γάμο και ε, νομική κατάσταση τέκνων. περιορισμένα το πεδίο εφαρμογής. Πολύ γλώσσα έντυπα θα υπάρχουν για ορισμένες περιπτώσεις, αλλά δεν θα είναι αυθύπαρκτα θα αποτελούν μόνο ένα βοήθημα για τη μετάφραση. Δεν θα υπάρχουν ως αυτόνομα έγγραφα που θα κυκλοφορούν παράλληλα με τα εθνικά έντυπα. Τα κράτη-μέλη δεν δέχθηκαν να υπάρχουν έντυπα διαφορετικά από τα εθνικά τους. Ε, σε σχέση με τη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών, διατηρείται το σύστημα ΙΜΗ τη ε, ανταλλαγή πληροφοριών ε, για την εσωτερική αγορά και μέσα σε πέντε χρόνια το Συμβούλιο προβλέπει την αναθεώρηση, δηλαδή τη μελέτη τη λειτουργία του συστήματο και τη ανταλλαγή τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών. Οι θέσει λοιπόν του Συμβουλίου απέχουν σημαντικά από αυτέ τι πρώτε ανάγνωση του Κοινοβουλίου και όμω αποτελούν ένα πρώτο βήμα για την απλούστευση της αποδοχής εγγράφων. Πρέπει να σημειώσω, να υπογραμμίσω ότι δεν πρόκειται για αναγνώριση εντύπων, αλλά για αποδοχή. Δεν γίνεται αυτόματα αμοιβαία αναγνώριση, απλώς γίνεται δεκτό ως αυθεντικό ένα έγγραφο και άρα μπορεί να το δεχθεί και να το χρησιμοποιήσει μια εθνική αρχή. Αύριο γίνεται πρώτος τριμερής διάλογος όπου θα γίνει η αξιολόγηση της κατάστασης και των αποκλήσεων των θέσεων για να καταλήξουμε σε χρονοδιάγραμμα που θα μας επιτρέψει να προχωρήσουμε στις συζητήσεις. Πιστεύω ότι χρήσιμο θα είναι καταρχάς να ακούσουμε τι έχουν να πούν οι σκιώδεις, οι συγητές για το θέμα αυτό και δεύτερο να προβλέψουμε για το περαιτέρω διάστημα μια συζήτηση με τους σκιώδεις συγητές ώστε να πούμε στις τρεις λεπτομέρειες άπαξ και λάβουμε τις λεπτομερείς θέσεις του Συμβουλίου. Αυτά είμαι στη διάθεσή σας και περιμένω ακούω τις θέσεις σας. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ζητάει κάποιος το λόγο. Ο κ. Ράντιεφ. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρο. Συνάδελφοι, όπως τα γνωρίζετε, τον Ιούνιο το Συμβούλιο κατέληξε σε μια γενική προσέγγιση όσον αφορά την απλούστευση αναγνωρίσεως κάποιων επισήμων εγγράφων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως οι πολίτες τώρα που πηγαίνουν σε άλλο κράτος μέλος ξοδεύουν και χρόνο και χρήμα για να αποδείξουν την αυθεντικότητα των εγγράφων τους ούτως ώστε να ε, βάλουν τη σφαγίδα της Χάγης ή να πιστοποιήσουν μια μετάφραση. Είναι ένα βήμα προόδου η θέση του Συμβουλίου, αλλά μείωσε το πεδίο εφαρμογή του κανονισμού του Συμβούλιο και εξαιρούνται πάρα πολλά έγγραφα που το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήθελαν να απελευθερωθούν από αυτές τις τυπικές διαδικασίες. Αυτό υπονόμευσε σοβαρά τα αποτελέσματα τα επιδιωκόμενα. Για να αρθούν οι γλωσσικοί φραγμοί, το Συμβούλιο προέβλεψε την ύπαρξη διαφόρων εντύπων ε, πολύγλωσσων σε όλες τις γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να μην χρειάζονται οι μεταφράσεις από τα 12 έγγραφα όμως που εκαλύπτονται από το πεδίο του κανονισμού μόνο τέσσερα θα καλύπτονται από τα πολύγλωσσα αυτά έντυπα. Ελπίζουμε να αλλάξει. Δοθέντος του χρόνου που απαιτήθηκε για να καταλήξει γενική προσέγγιση στο Συμβούλιο Νομίζω ότι μας περιμένουν σκληρές διαπραγματεύσεις στον τριμερή διάλογο. Ελπίζω ότι με, τον εισηγή... με την εισηγήτρια και τους κοιόδης θα προχωρήσουμε και έτσι θα διευκολύνουμε την καθημερινή ζωή των πολιτών αντί να την περιπλέκουμε. Αυτά και ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ πολύ. Ζητά κάποιος άλλος το λόγο μήπως. Ήταν πολύ σύντομη ανταλλαγή απόψεων. Αυτό θα έλεγα εγώ. Εάν πράγματι περί αυτού πρόκειται, η κυρία Ντελφό θέλει να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ ακόμα και για τη σύντομη αυτή ανταλλαγή των απόψεων. Συνεπέρανα ότι μπορούμε να προχωρήσουμε στις διαπραγματεύσεις και θα καλέσω τους σκιώδεις το Σεπτέμβριο για να συζητήσουμε το θέμα λεπτομερέστερα. Να επενθυμίσω ότι το απόγευμα ο Λουξεμβούργος Υπουργός ο Κεσμπραντς θα παρίσταται και μπορούμε να του θέσουμε ερωτήσεις και επ' αυτού. Από ό,τι κατάλαβα, η Προεδρία θα παρέμβει τώρα το απόγευμα. Ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες. Πράγματι δεν ζητεί κάποιος άλλος τον λόγο. Εξαντλήσαμε το πρωινό μας πρόγραμμα, οπότε σας εύχομαι καλή σας όρεξη και γεια σας.